ανάμεσά μας μία αντιπροσωπεία του Γεωργιανού Κοινοβουλίου με την πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Uh, which just took place. I'm particularly happy to welcome you in our plenary, especially on this occasion, and I'm certain that you have had Είμαι βέβαιος ότι οι συζητήσεις τις οποίες είχαμε όλοι με τους αντιπροσώπους του Κοινοβουλίου της Τυφλίδας ήταν παραγωγικές. Διακόπτουμε και θα ξεκινήσουμε σε λίγα λεπτά με την ομιλία του Πρωθυπουργού του Καναδά.